Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Είναι Δευτέρα, είμαστε Στρασβούργο και θα ξεκινήσουμε αρχικά εγκρίνοντας το σχέδιο μερικές διάταξης. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Η διερμηνία είναι σε 19 γλώσσες διαθέσιμη. Θέλω να σας πω ότι στις 20 Ιουνίου η Επιτροπή μας αποφάσισε για να γνωμοδοτήσει για το σώμα αλληλεγγύης. Με βάση το νέο άρθρο 53-4 του κανονισμού. και η αρμόδια καθήλυνη Επιτροπή Πολιτισμού τη θέση της αντιπαρουσιάσης από τη μορφή τροπολογιών. Εμείς έχουμε βάλει προθεσμή για την κατάσταση τροπολογιών την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Μέσω του συστήματος AT4AM ε, και ψηφίζουμε στις 6 Νοεμβρίου. Το επόμενο σημείο ο κύριο Χόισλινγκ έχει ζητήσει το λόγο, αλλά πάρα πολύ γρήγορα παρακαλώ. Στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε ό,τι αφορά το σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη, ε, που είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ε, ενέργεια, να το αναβάλουμε, να μην το ψηφίσουμε απόψε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαδικασία, το έγραψε και η συγκήτρια θα ήταν ε, καλό να μην γίνονται ε, συναντήσεις ε, όπου θα αποφασίζονται συμβιβαστικές προτάσεις με την απουσία όλων των σκιωδών συγκητών. Δεν είναι δυνατόν. Η Περιβάλλοντος έχει αναβάλει για τα τέλη Οκτωβρίου την ψηφοφορία. Επομένω και εμεί έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε με τι ομάδε και να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη τελική πρόταση. Έλα, επομένω ζητώ αναβολή του σημείου 5 για την επόμενη φορά. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα ω Επιτροπή Γεωργία, πιστεύω. Ο πρόεδρος, με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει από τη γραμματεία, δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμη για το κατά πόσον θα αναβληθεί πράγματι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος η ψηφοφορία. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό ακόμη στην Επιτροπή. Ενδύ... Εσείς. Η κυρία Πετήρ. Επειδή, συνάδελφοι, εγώ δεν συμφωνώ με το έτοιμο του κυρίου Χόισλινγκ περί αναβολής ψηφοφορίας, διότι έχουμε κάνει πολύ δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις και έχουμε καταλήξει σε συμβαστικές προτάσεις των οποίων συμφωνούν περισσότερες πολιτικές ομάδες. Έγιναν τέσσερις συνεδριάσεις και οδών εισηγητών, υπήρξαν και άλλες τρεις τεχνικές συναντήσεις. Προσωπικά εγώ έχω συζητήσει με τους περισσότερους από τους σκιώδεις εισηγητές και μάλιστα επανειλημμένους για να κατανοήσω τη δική τους θέση και με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτική η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Είναι σημαντικό, νομίζω, να εγκρίνουμε μια ξεκάθαρη γνωμοδότηση πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, που πολύ σωστά είπατε, δεν έχει αποφασίσει ακόμη αναβολή τη ψηφοφορία. Άρα δεν είναι σωστό αυτό. εμείς. εδώ είμαστε για να υπηρετήσουμε τους αγρότες, τα δικά του συμφέροντα και για να επιβιώσει και να ανθίσει η γεωργική ε, ύπεθρος γεωργικές περιοχές. Γι' αυτό ζητώ λοιπόν να μην αναβληθεί το σημείο και να ψηφίσουμε. Πρόεδρος. Ακούσαμε τις απόψεις. Μίλησε και η συγγήτρια. Όποιος θέλει το λόγο, πολύ σύντομα παρακαλώ. Κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ πολύ. Δι... Ε, σπάνια συμβαίνει να υποστηρίξω τον Μάρτιν Χοσλίνκ, αλλά εγώ θέλω να καθυστερώ την νομοθεσία στο σώμα, ιδίω δε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπω είναι η ενέργεια. Είμαι στο πλευρό του για αυτή τη φορά, γιατί αυτό είναι ο ρόλο μου, να καθυστερώ την νομοθεσία. Να μην χάσουμε χρόνο όμως. Ποιον βοηθάτε πιο πολύ δεν ξέρω με αυτά που είπατε βέβαια την εισηγήτρια ή τους Κιώδης, ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η του κιωδης ο κύριο τακουλα έχει κάνει Κύριε δουλειά. Υπήρξε υπομονετική μαζί μας με τους Κιώδης εισηγητές. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω πλήρως ε, τη δουλειά που έχει κάνει και δεν καταλαβαίνω την άποψη Χόισλινγκ Εγώ λοιπόν είμαι στο πλευρό της κυρίας Πετήρ, γιατί νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως εισηγήτρια και μας άκουσε τους Κιώδης. Πρόεδρος. Κύριος Αντριέ, να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταλαβαίνω πλήρως το αίτημα του κυρίου Χάουσλινγκ, επειδή είναι σημαντική αυτή η νομοδότηση, Πρόοδο κάναμε, ε, προχωρήσαμε, ε, το είπε και η κυρία Πετήρ, και παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμη επεξεργασία η έκθεση ε, για την ενέργεια και το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει συνένεση. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, πιστεύω, εντελώς το έργο μας. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της αναβολής, όπως ζήτησε ο κ. Χόισλινγκ. Ευχαριστώ, κυρία Σένρα. Ευχαριστώ. Εγώ με την πλευρά μου, από την πλευρά μου θέλω να υποστηρίξω την πρόταση του κυρίου Χόισλινγκ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Προτείνω λοιπόν. Α, ο κύριο Νταντά. έχω μείνει έκπληκτος με αυτά που ακούω. Δεν είμαστε καν βέβαιοι ότι δεν θα ψηφίσει τι επόμενες ώρες η Ένβη. Και εμείς να κινδυνεύουμε, παίρνουμε ένα ρίσκο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα να μην έχουμε γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας. Τι κάνουμε με τις ευθύνες μας. Δομάδες είχαμε στη θέση μας για να προετοιμάσουμε την έκθεση αυτή. Είναι δύσκολη, λυπούμε, αλλά δεν ήταν η μόνη. Έχουμε συστήσει πολλέ τέτοιε δύσκολε εκθέσει στην Επιτροπή μα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εμεί δεν θα έχουμε αποφανθεί πριν την Επιτροπή Περιβάλλοντο. Πρόεδρος. Ζήτησα πριν από λίγο από τον υπεύθυνο της γραμματείας, της γραμματείας να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο για το κατά πόσο θα αναβάλει η ΕΝΒΗ την ε, ψηφοφορία. Και αν δεν το κάνει, ε, που δεν έχουμε κάποιο τέτοιο νέο, εμείς δεν θα μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε. Καταλαβαίνω ε, και άκουσα όλους όσου ήθελαν το λόγο. Οπότε τώρα προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του αιτήματο Χόισλινγκ. Ηλεκτρονικά βέβαια θα ψηφίσουμε, έτσι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την πρόταση Χόισλινγκ. E Ένα από το ΕΛΚ παραπάνω. Πρέπει να βγάλει κάποιο ο υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Εντάξει, λύθηκε το θέμα. Το Εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία κάθε αυτή για, ως προς τη συστάσεις σε σχέση με την εντολή διαπραγμάτευσης για την Αυστραλία η γνωμοδότηση, ε, ο εισηγητής με συγχωρείτε είναι ο κύριος ε, Άντριε. Η Ίντα Κομίτη είναι η επικεφαλής και όπως θα γνωρίζετε έπρεπε να εργαστούμε τάχιστα για αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Αντρίο θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι οι δύο ε, κοινέ εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές για τον τομέα της ε, γεωργίας. Κάναμε μια πολύ καλή συλλογική εργασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που προέβαλαν τροπολογίες ιδιαίτερα χρήσιμες. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε μια, σε μια συνενετική στάση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία που μας βοήθησε στην όλη εργασία. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις συμβαστικές. Ε, ε, ένα, τροπολογία ένα, υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Δύο, υπέρ σας ευχαριστώ, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε εφόσον το επιθυμείτε. 22. Αρχίζει ο έλεγχος για την 22. Ένας ε, σοσιαλιστής υπεράριθμος, παρακαλώ να αποσύρει την κάρτα του. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. 39 παρακαλώ. Υπέρ υπέρ εγκρίνεται. 40 υπέρ εγκρίνεται. 55 υπέρ εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά απορρίπτεται. 58 υπέρ εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά απορρίπτεται. 65 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Ευχαριστώ εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 118 υπέρ, εγκρίνεται. 100 υπέρ, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Αλλά θα ελέγξουμε. 108 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. 109 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Κατά λίγες ψήφους. 112 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά απορρίπτεται 115 υπέρ κατά ελέγχουμε 115 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται 117 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε τώρα το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί. Η ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε και εγκρίνεται συγχαρητήρια. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ εντάχει. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη σύμπνοια και πιστεύω ότι η πρόταση είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Έτσι ε, αποστέλουμε ένα θετικό πρόσημο σε σχέση με αυτό τον ένα αγώνα υπέρ των ελευθέρων συναλλαγών. Στο τομέα της γεωργίας. Θέλουμε εμείς να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των συμφωνιών που επιτυγχάνονται σε επίπεδο, στο επίπεδο του τομέα μας. Εξαιρετικά η προετοιμασία αυτής της γνωμοδότησης. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Από ό,τι κατάλαβα, ο εισηγητής θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις ε, και αν υπάρξουν θέματα ε, για τα οποία θα πρέπει να μας ενημερώσετε, θα ήθελα να σας ζητήσω να παρέμβετε και να φροντίσετε να μας γνωστοποιηθούν, ε, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια λεπτά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η αρμόδια επί επιτροπή είναι η Επιτροπή Ίντα, υπενθυμίζω. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, ε, γνωμοδότηση για τη διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία. Και πάλι η αρμόδια επί της επιτροπή είναι η Επιτροπή Ίντα. Και ο κύριος Κασπαρή ε, είναι ο εισηγητής ε, για την Επιτροπή Ίντα και ο κύριος Νίκολσον είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ο κύριε Νίκολσον, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχανε. Έρχεται σε μια δύσκολη και αρκετά ε, λεπτή στιγμή για μας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και επομένως ε, θα πρέπει να ευχαριστήσω όχι μόνο το προσωπικό της γραμματείας ε, αλλά και το προσωπικό μου στο ομάδα, το ECR και τους κοιόδης συγητές οι οποίοι συνεργάστηκαν πολύ καλά μαζί μου και τους ευχαριστώ διότι καταλήξαμε σε μια πολύ ισορροπημένη γνωμοδότηση και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα γιατί έχουμε και αρκετή δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι μετά την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία ή μάλλον τροπολογία 4. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ή μάλλον συγγνώμη, ήθελα να πω συμβιβασμό, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβασμό Α. πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στη συμβαστική τροπολογία B1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε Στην τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική C. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία E. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή, τον κύριο Αντριέ και τους κυρίους Δενανό και Μέκοφ. Έχω την έγκρισή τους και προτείνω μια ε, προφορική τροπολογία για να συμπεριλάβουμε δύο φράσεις τις οποίες θα διαβάσω στα αγγλικά. Μετά, after those sectors. Especially with regards to the monopolistic structure of some industries, and in particular of the dairy sector in New Zealand. Και μετά συνεχίζει η τροπολογία ως έχει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Γκρίνεται λοιπόν η προφορική τροπολογία και ε, ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Να κάνουμε όμως μια παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 67. Θα έλεγα βέβαια ότι εγκρίνεται. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 68. Υπέρ. Κατά. Μια σύγχυση βλέπω στα μέλη του ΕΛΚ. Επαλήθευση λοιπόν για την 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 68. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 69. Πέρα εγκρίνεται. 70. Δεν υπάρχει ψηφοφορία, είναι γλωσσικό. Συμβιβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά απορρίπτεται 82 υπέρ κατά απορρίπτεται Ογδόντα έξι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. 90 υπέρ. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 101 υπέρ, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 108 υπέρ, Να κάνουμε μια επαλήθευση. Για την 108. Άρχεται η ψηφοφορία. 108. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, αλλά με μικρή διαφορά. 112 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά επαλήθευση για την 111 άργια την ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 113 υπέρ κατά απορρίπτεται 116 υπέρ κατά απορρίπτεται 118 υπέρ κατά Απορρίπτεται, αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση για την 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής θέλει και πάλι το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Συγχαρητήρια. Και να συγχαρώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω και εσάς να συνεχίσετε να παρακολουθείτε την ε, εξέλιξη των εργασιών για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Στις 12 Οκτωβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Ίντα. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα θα ή μάλλον αν δεν υπάρχει πρόβλημα θα συζητηθούν όλα στην επόμενη ολομέλεια. Τώρα, ε, προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ε, η κυρία Πετήρη είναι η συγκήτρια για τη γνωμοδότηση αυτή. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για την Επιτροπή μας. Δύο είναι οι αρμόδιες επιτροπές, η Άγκρη και η Τραν. Η Τραν έχει ζητήσει τη συμμετοχή μας βάσει και του άρθρου 53 το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε και ο ίδιος είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δύσκολο, βαρύ και είμαι ικανοποιημένη διότι με τις περισσότερες πολιτικές ομάδες ε, κατάφερα να καταλήξω σε καλές συμβαστικές προτάσεις και πιστεύω ότι μετά την έγκριση της ε, νομοδότησης θα έχουμε μια σαφή θέση ως Επιτροπή Γεωργίας. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές, τους βοηθούς, συνεργάτες τους για τη βοήθειά τους. Διότι πιστεύω ότι τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Ιδιαίτερος θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Βασίλη που βοήθησε ε, από τη γραμματεία. Είχαμε καιρά τη λίστα σοφορείο Να ευχαριστήσω και τη βοηθό μου και τον κύριο Strange και ζητώ από όλους τους ε, συναδέλφους μου να στηρίξουν την εκτίμηση. Είναι πολύ σημαντική για το περιφάλλον το αγροτικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Ο πρόεδρος, όπως είπα, είναι δύσκολο το θέμα. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα, αλλά τελικά τα επιλύσαμε. Ας ξεχάσουμε λοιπόν το παρελθόν και να ψηφίσουμε τώρα την έκθεση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 223 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 224, 25, 26 από κοινού είναι ταυτόσιμες παρόμοιες τέλο πάντων υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκαν. 227 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε, λυπούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Δεν το βλέπα. Τέσσερι μόνο ψήφισαν. 228 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 229 ε, υπέρ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 και 230. Γίνεται ταυτόσιμες υπέρ. Εγκρίνονται. 232 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 233 υπέρ, εγκρίνεται. 234 υπέρ, εγκρίνεται. 235, 36, 37 υπέρ, εγκρίνεται. Εντάξει, θέλετε να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία πέρας. Άρα μπορώ να πω ναι, μπορώ να πω και όχι. Ισοψηφία. Άρα να που δεν απορρίπτονται πάντα οι προτάσεις μικρότερων ομάδων. 238 ψήφι υπέρ. Κατά. Ε, γκρίνεται, όχι, ας επαληθεύσουμε, ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά, εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 240 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Εντάξει, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 241-42 μαζί. Είναι παρόμοιες ψήφοι υπέρ. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 245 τώρα. Ψήφι υπέρ. 245 είπα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. την 247 και 248 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 254 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Τη 254 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 200 55 τώρα ψήφι πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 και 258-259 μαζί. Ψήφι πέρ Εγκρίνονται. 261 υπέρ. Εγκρίνεται. 263. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 264. Υπέρ. Εγκρίνεται. 266 και 67. Ψήφι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Όχι. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 2.75 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2.76 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 292 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 294. 294, τι κάνουμε, ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ, Λοιπόν, 2.94 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Τη 2.94 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 17. Τρεις σελίδες μετά. Μαζί με την 321 ταυτόσιμες ψήφι πέρ. Κατά. Φαίνεται να έχουν απορριφθεί, αλλά σε ελέγξουμε. Τις τροπολογίες 17 και 321. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίστε. Αφού μιλάτε εκεί πέρα. Πέρασε φοβορίας. Με μία ψήφο διαφορά απορρίφθηκαν. Πού πηγαίνουμε. Στην 322 ψήφι πέρα. Κατά. Απορρίπτεται. 328 ψήφι περ. Κατά. Απορρίπτεται. 323 ψήφι περ. Κατά. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Εγκρίνεται. 325 ψήφι περ. Κατά απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 327 ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 333 ψήφι υπέρ, κατά εγκρίνεται. 335 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 336 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 337 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 338 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 339 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 340 υπέρ, κατά απορρίπτεται 341 υπέρ κατά απορρίπτεται 342 υπέρ κατά απορρίπτεται 343 υπέρ κατά απορρίπτεται 344 υπέρ εγκρίνεται 345 υπέρ κατά απορρίπτεται 346 υπέρ Εγκρίνεται. 347 υπέρ. Εγκρίνεται. 348 υπέρ. Εγκρίνεται. 349. Θέλετε να ελέξουμε την 348. Εντάξει, ξεκινάει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 349 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 350 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 351 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 352 υπέρ, εγκρίνεται. 353 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 354 υπέρ, εγκρίνεται. 355 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 356. Εντάξει, εντάξει. Ελέγχουμε 355. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 356 υπέρ κατά απορρίπτεται. 357 υπέρ εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά απορρίπτεται. 359 υπέρ κατά απορρίπτεται. 360 υπέρ κατά απορρίπτεται. 361 υπέρ κατά απορρίπτεται. 362 υπέρ κατά απορρίπτεται. 363 υπέρ εγκρίνεται 364 υπέρ, κατά απορρίπτεται 365 υπέρ, εγκρίνεται 366 υπέρ, κατά απορρίπτεται 367 υπέρ, κατά απορρίπτεται 368 υπέρ, κατά απορρίπτεται 369 υπέρ, κατά απορρίπτεται 370 υπέρ, κατά απορρίπτεται 371 υπέρ κατά απορρίπτεται 372 υπέρ εγκρίνεται ελέγχουμε ελέγχουμε 372 άρχεται η ψηφοφορία βλέπω ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ πέρας Απορρίπτεται. 373. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 375 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 375 άρχεται η ψηφοφορία. Ίσως προχωρά πολύ γρήγορα για μερικούς. Πέρας. Απορρίπτεται συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Κανένα σχόλιο λέει ο πρόεδρος. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 410. 410 εγκρίνεται. 24 υπέρ. Εγκρίνεται. 411 εγκρίνεται. 412 εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 414. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 415 και 16 εγκρίνονται. 417 υπέρ εγκρίνεται. 418 υπέρ εγκρίνεται. 419 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 445. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 441 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 430 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 431, 32, 33 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 438 υπέρ κατά απορρίπτεται 439 για 440 από κοινού υπέρ κατά απορρίπτονται συμβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 472 ε, περνάμε τρεις σελίδες, 472. Τη βρήκατε? Υπέρ. 472 υπέρ, ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 471. άμε συγχωρείτε, έκανα λάθος μάλλον. 400 74. Υπέρ. Εγκρίνεται. 475 υπέρ. Εγκρίνεται. 473 υπέρ. Εγκρίνεται. 476 υπέρ. Εγκρίνεται. 478 υπέρ κατά απορρίπτεται. 479 υπέρ κατά απορρίπτεται. 480 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 494. 494 υπέρ Κατά. Θα ελέγξουμε. 494. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 501 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε. Αφού το θέλετε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 502 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 503 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε. 503 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 504 υπέρ. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 504. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 508 υπέρ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 510 υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 510. Πέρας. Απορρίπτεται. 511 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 512 υπέρ, εγκρίνεται. 40 υπέρ, εγκρίνεται. 41 υπέρ, εγκρίνεται.

521 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 520-522 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Θα ελέγξουμε τις δύο τροπολογίες αυτές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 523 υπέρ, 523 υπέρ εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά εγκρίνεται. 63 υπέρ εγκρίνεται. 64 υπέρ εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 66 υπέρ, εγκρίνεται. 67 και 68 υπέρ, εγκρίνονται. 69 και 70 υπέρ, εγκρίνονται. 71-72 υπέρ, εγκρίνονται. 76 υπέρ. Για άλλη μια φορά παρακαλώ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 78 και 79 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 80 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 81 υπέρ, Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οι 86 και 87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 88 και 89 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Να κάνουμε όμως μια επαλήθευση. 88 και 89. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. απορρίπτονται. Έχει τόσο πολλά επίθετα εδώ που πραγματικά δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. 90. Εγκρίνεται. 91 και 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Απορρίπτονται, συγγνώμη, 93. Επαλήθευση για τις 91 και 92. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 93 υπέρ. Κατα... 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 110-111 υπέρ, εγκρίνεται. 112 υπέρ, Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση. Ωραία. 110-111. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι εκρίνονται. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Δεν ε, σχολιάζω. 112 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Α. Ε, εγκρίθηκε 115. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. για την 117 εγκρίνεται. Η 99 εγκρίθηκε. Πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία για την 101. Ε, Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Είμαστε τώρα στην 117. yeah, here, Sorry. 115. 115. 115 była odrzucona. Jesteśmy przy... Η 115 απορρίφθηκε. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για το 116. 115 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 117 είναι εξαιρετική, λέει ο κύριο Ταραμπέλα, πολύ καλύτερη από τη συμβαστική τροπολογία 1, επομένω έγινε δεκτά. Επομένω η 117, 118, 119 καταπίπτουν. Και πρέπει να πάμε στην 120. Ναι, αλλά ήμασταν στην 120, στην 116, συγγνώμη. Και μετά από την 116 θα πάμε στην 120. 120 λοιπόν τώρα, υπέρ. Υπέρ της 120, κατά απορρίπτεται. 121, 122, 123, υπέρ, κατά, να επαληθεύσουμε. 121, 122, 123. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 124, 125, 126 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 127 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 130 υπέρ, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά απορρίπτεται. 134 υπέρ εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά απορρίπτεται. 136 επαλήθευση. Ε, άρχεται η ψηφοφορία για την 136. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά εγκρίνεται 143 υπέρ κατά επαλήθευση ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 164 περνάμε. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Σκοτ υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 165 υπέρ, εγκρίνεται. 166 υπέρ, εγκρίν, κατά, απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, Ψηφίζουμε πρώτα την 167. 167 υπέρ. Κατά. Συνάδελφοι, ψηφίζουμε την 167. Μόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί θα αποφασίσουμε. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην 169. 169 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 178. 178, υπέρ, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 181 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 184 υπέρ, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Επαλήθευση όμως για την 186. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση για την 190. 190 πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 193 194, συγγνώμη, υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 194, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 203 υπέρ εγκρίνεται. 215. 215 υπέρ. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Εγκρίνεται. 217 υπέρ. Εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 219 υπέρ. Εγκρίνεται. 220. Ο κύριος Άγνιου έχει ζητήσει επαλήθευση. Γιατί 220 υπέρ κατά απορρίπτεται. 200 24 υπέρ κατά 524, 525 υπέρ, κατά 526 υπέρ εγκρίνεται, 527, 28, 29, 30 υπέρ εγκρίνονται. 531 υπέρ εγκρίνεται, 532 υπέρ εγκρίνεται, 533 υπέρ εγκρίνεται, 534 υπέρ εγκρίνεται, 536 υπέρ εγκρίνεται, 537 υπέρ εγκρίνεται. 538-539 υπέρ εγκρίνονται. Συγχαρητήρια στον κύριο Σάνι, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία 10. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Πέραση τη πληροφορία. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 10. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Πετήρ. Θέλετε τον λόγο? Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υποστήριξαν αυτήν την έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη ως Επιτροπή Γεωργίας ότι αφορά τη βιομάζα και τις ανανεώσιμες πηγές εν γέννη. Ελπίζω και οι Επιτροπές ΕΝΒΙΝΤΑ θα λάβουν υπόψη ε, τις ε, δικές μας απόψεις. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν ε, μάλλον έχουν σχετιστεί με τη γεωργική παραγωγή τα τελευταία χρόνια και με συζητήματα δασοκομικά η δασοκομεία, η γεωργία επηρεάζουν το περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει συνέργειες πολιτικές, ώστε οι τιμές να είναι προσιτές, αλλά και η ενέργεια να διατηρείται. Και θέλουμε να είμαστε και αυτά και στην παραγωγή πρωτεϊνών για τις οτροφές. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, στην Ήπεθρο. Η έκθεση αυτή λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν όπως επίσης τη Γραμματεία και, τις πολιτικές μας ομάδες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και τους και και όλους τους υπόλοιπους. Και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, προσοχή ε, στην ατμόσφαιρα. Ε, γιατί κάποιες φορές για λίγα πράγματα ασήμαντα μπορεί να έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ μας. Καλό είναι λοιπόν να τα βρούμε σε ένα καφέ και τα λοιπά, να προσέχουμε την ατμόσφαιρα και τις σχέσεις μας. Και ευχαριστεί ο πρόεδρος και τους διερμηνείς. Επόμενη συνεδρίαση 9, 10 και 11 Οκτωβρίου και στις 11 Οκτωβρίου Επιτροπή ΕΝΒ και εμείς κοινή συνεδρίαση, δημόσια ακρόαση.